Όχι, τα πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται. Θα ήθελα τώρα να σας ανακοινώσω πως σήμερα το πρωί επέστρεψα από επίσημη επίσκεψη στην Ρωσία. Η πρώτη επίσκεψη Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ και 12 χρόνια. Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο Μετβέντεφ, τον Πρόεδρο της Δούμας Μπόρις Γκρίσλοφ, του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ρεσκέη Γκρίσλοφ και τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ενέργειας. Μιλήσαμε για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένωσης-Ρωσία στο πλαίσιο της συνεργασίας για τον εξυγχρονισμό και την πιθανότητα νέας συμφωνίας ε, διμερούς. Ε, συζητήσαμε και άλλα ζητήματα, μεταξύ των οποίων το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης συναντήθηκα με εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας ε, των πολιτών, μεταξύ των οποίων και της οργάνωσης Memorial που έλαβε το βραβείο Ζαχάροφ το 2009. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου κλιμακώθηκε η διαφωνία με τη Λευκορωσία για το φυσικό αέριο. Διαβίβασα την ανησυχία μας στις ρωσικές αρχές και ζήτησα από τα δύο μέρη να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις για την παράδοση φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης σημείωσα πως ε, θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές ρήτρε στις συμβάσει μεταξύ Λευκορωσίας και Ρωσίας που θα εγγυώνται την παροχή αερίου στην Ένωση. Η, η εγγύηση αυτή είναι το σημαντικότερο για εμάς. Επίσης, Κομισιόν και Συμβούλιο εξετάζουν το ζήτημα. εσείς, λοιπόν οι πρόσωποι μπορούσαν να μας ενημερώσουν κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση αλλάζει, βρίσκεται εν εξελίξη, κάθε ώρα έχουμε νέες πληροφορίες σε σχέση με αυτή